Επίσης να σας πω ότι λίγη η σημερινή συνεδρίαση και η επόμενη θα είναι αύριο το πρωί με την ημερήσια διάταξη η οποία έχει δημοσιευθεί και στο έγγραφο της συνεδρίασης αλλά και στο ίντρανετ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλό βράδυ. Τέλος συνεδρίασης.